Nous Καλώς, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και έχουμε τη χαρά να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων σήμερα το απόγευμα με τον κύριο Μάρκο Πάβιτς, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω. Είστε Υπουργό Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ευρωπαϊκών Ταμείων. Είστε ασκόν την Προεδρία του Συμβουλίου. Σχετικά, θα μα μιλήσετε σχετικά με τι προτεραιότητε τη Κροατική Προεδρία. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μα που σα υποδεχόμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ, σήμερα το απόγευμα για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εξή επόμενοι μήνε θα είναι μήνε εντατική εργασία και θα είναι μήνες καθοριστικοί για τη λήψη των αποφάσεων αναλαμβάνετε την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια χρονική στιγμή που αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική ε, συγκυρία. Διότι πρέπει να ξεκινήσει ξανά η διαπραγμάτευση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τη στιγμή κατά την οποία η Φιλανδική Προεδρία έχει καταθέσει μια πρόταση η οποία γνωρίζεται ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αποδεκτή. Είναι μια πρόταση την οποία εμείς απορρίπτουμε, την οποία εμείς αρνούμαστε και ως προς το συνολικό προϋπολογισμό που προτείνεται και ως προς τις πτώσεις και τις μειώσεις και τις περικοπές ε, των χρημάτων που δίδονται σε ορισμένες πολιτικές και πιο συγκεκριμένα την πολιτική της συνοχής που μας αφορά εμάς εδώ στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή και θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά όταν έχουμε νέους στόχους και όταν θέτουμε νέους στόχους πρέπει να έχουμε νέα μέσα και νέα ταμεία και νέα κονδύλια τα, οι νέοι στόχοι που έχουν ε, οριστεί είναι πολύ άριθμοι, όμως τα κονδύλια και τα ταμεία που προβλέπονται, το μόνο που κάνουν ε, είναι να οπισθοχωρούν σε ό,τι έχει να κάνει με το μέγεθος και τον όγκο τους. Θα τα πούμε όλα αυτά, το ίδιο όμως ισχύει από πλευράς μας και για τη μέθοδο διαπραγμάτευσης. Έχουμε το περιβόητο κοιτίο διαπραγμάτευσης, negotiative box μάθαμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και ε, αυτό δεν σέβεται τους κανόνες και τις αρχές της συναπόφασης. Δεν σέβεται τις αρχές της συναπόφασης έτσι όπως ε, διατυπώνονται στις συνθήκες. Το Συμβούλιο ε, τρόπον την υπερβαίνει των αρμοδιοτήτων του και έρχεται να επικαλύψει νομοθετικές αρμοδιότητες ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τα κείμενα και τις ε, συνθήκες. Επομένως, στηρίζουμε πλήρως την απόφαση που υιοθετήθηκε στις 19 του περασμένου ε, Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, την απόφαση από τη διάσκεψη των Προέδρων και γι' αυτό οι συντονιστές μας στη συνεδρίασή του σήμερα το πρωί έλαβαν την εξή απόφαση για την Επιτροπή ΡΕΤΖΙ Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα παγώσουμε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου τον τριμερή πολιτικό διάλογο ε, τον καταληκτικό. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν να παγώσουμε τον ε, τριμερή πολιτικό διάλογο, τον τρίλογο αυτό δηλαδή. Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει κάτι το οποίο αποτελεί και δική μας βούληση. Δηλαδή να συνεχίσουμε να προχωρούμε, να σημειώνουμε πρόοδο με την Κροατική Προετία σε συνεδριάσεις τεχνικού ενδιαφέροντος και γιατί όχι και σε συνεδριάσεις με άλλη μορφή για να σημειώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο και έτσι ώστε να μπορούν οι περιφέρειες μέσα στις προσήκουσες προθεσμίες να έχουν κανονισμούς που να ρυθμίζουν τη χρηματοδότησή τους. Προετοιμαζόμαστε όμως για όλα τα ενδεχόμενα και για όλες τις επιλογές, διότι δεν μπορούμε με πρόσχημα τη βιασύνη να δεχθούμε το οτιδήποτε και το ό,τι να είναι. Περιμένουμε λοιπόν από το Συμβούλιο να ε, καταθέσει πρόταση για προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι στο, στο ύψος των προκλήσεων που μας επιβάλλει ο στόχος της συνοχής. Και περιμένουμε από το Συμβούλιο να καθορίσει ε, την άποψή του για το σύνολο των άρθρων που άπτονται των κανονισμών που αποτελούν αρμοδιότητά μας να διαπραγματευτούμε και που δεν αποτελούν μέρος του κοιτίου διαπραγμάτευσης όπως σας το ανέφερα. Σήμερα το πρωί είχαμε μακροσκελή, μακροσκελή ε, εις βάθος συζήτηση με την Επίτροπο Αρμόδια Ελίζα Φερέιρα και μιλήσαμε αρκετά για το μηχανισμό της δίκαιης μετάβασης και θα πρέπει να ε, δουλέψουμε σε αυτό το μηχανισμό μαζί σας, πάνω σε αυτό το μηχανισμό και περιμένουμε τη θέση σας ε, για αυτά τα ζητήματα. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν μπορείτε εσείς να μας πείτε το, το πόσο πρόκειται να προχωρήσει για το θέμα αυτό η Προεδρία σας. Ποια, ε, ποιο είναι το όραμα της Προεδρίας σας για αυτό το μηχανισμό και για τη διαιτησία ε, έτσι όπως προβλέπετε στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μας Επιτροπή θα ολοκληρώσει το νομοθετικό της έργο, την νομοθετική της πρωτοβουλία και στο τέλος όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα μάθετε τη θέση της Επιτροπής Ρέτζη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου αυτής της χρονιάς αναλαμβάνεται την Προεδρία. Στη συνέχεια θα πάρει, τα, ε, θα πάρει τη σκητάλη η Γερμανική Προεδρία από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Οι προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας παρα κατατίθενται στο έγγραφο της Προεδρίας, μια ισχυρή Ευρώπη, για αυτήν κάνετε λόγο. Έχετε μοιράσει το έγγραφο στο σύνολο των συναδέλφων και λέτε ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ισορροπημένη ανάπτυξη των περιφερειών. Είπατε ότι θα υπερασπιστείτε την πολιτική συνοχή στην οποία είπατε ότι θεωρείτε κρίσιμη σημασία. Και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας είπατε ότι θα οργανώσετε διάφορες επίσημες ή και άτυπες εκδηλώσεις για να ενισχύσετε την ορατότητα της περιφερειακής πολιτικής. Και οφείλω να σας πω ότι αυτά τα μελούμενα και αυτές τις ανακαινώσεις τις ακούμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. ευχαρίστηση. Το γεγονός ότι θα υπάρχει για παράδειγμα άτυπο συμβούλιο για θέματα συνοχής. Ε, αν δεν απατώμε ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Γενικών Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, το οποίο θα ασχοληθεί και με το θέμα της συνοχής. Επίσης θα σας ακούσουμε να μας παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τα ευρωπαϊκά νησιά και ότι σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα στο θέμα της νησιωτικής Ευρώπης. Και με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε τις προτάσεις σας για τα θέματα αυτά. Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να αναλάβετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για το θέμα των νησιών, ένα θέμα το οποίο είναι ε, προτεραιότητα στην ε, ε, ημερήσια διάταξη για το μέλλον. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σας υποδεχόμαστε εδώ. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές και μετά με τα μέλη της Επιτροπής σας δίνω το λόγο για να παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας και στη συνέχεια θα υπάρξει συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Poštovani predsjedatelju odbor, odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj, gospodine Omarži, poštovani zamjenici predsjedatelja, članovi odbora. i της Επιτροπής, Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας ε, ε, υπεύθυνος για περιφερειακά ζητήματα και διαρθρωτικά ταμεία. Για μένα είναι μεγάλη τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα προνομιακή αλλά και δύσκολη η θέση μου. Λέγομαι Μάρκο Πάβιτς και είμαι Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Κροατία. Το Υπουργείο μου είναι υπεύθυνο για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται ο Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων. Χαρτοφυλάκιο που είχα πριν από το παρόν. Άρα μπορώ να πω ότι έχω πείρα σε θέματα διαρθρωτικών ταμείων στην ε, Κροατία. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Ε, παλαιότερα, το 2014, ήμουνα και εγώ σταζιέρ. Ο Αντρέ Πλένκοβιτς ε, ήταν ο ευρωβουλευτής μου τότε, τώρα είναι πρωθυπουργός της Κροατίας. Το 2016 ασχολήθηκα με την πολιτική νεότητας και τα ευρωπαϊκά σχέδια για τους νέους στην αγορά εργασίας. 30 νέοι μπόρεσαν να βρουν θέσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επισκέφθηκαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δική μου πρωτοβουλία το 2016. Ε, κατέχω μάστερ που αφορά τις κλιματικές αλλαγές και φυσικά γνωρίζω πολύ καλά και το Πράσινο Σύμφωνο καθώς και τα χαρτοφυλάκια που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές καθώς και το ε, Ταμείο Μετάβασης. Όλα αυτά είναι, θα μπορούσα να πω, ενταγμένα στο DNA μου. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα από όλες τις απόψεις. Πιστεύω η Κροατία είναι το νεότερο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς να αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα εργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο αλλά θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Χωρίς διαφοροποίησης θέλουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι, δεχόμενοι τη διαφορετικότητά μας. Αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, όχι πολύ καιρό πριν ζήσαμε μια εμπόλεμη κατάσταση, αλλά καταφέραμε να ελευθερωθούμε και να ζούμε στην ελεύθερη Κροατία, η οποία είναι μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Όπως ξέρετε, η Κροατία ανήκει στον, στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, που είναι αναπόσπαστος λίθος για την ευημερία της. Έχουμε το, της το, τη μεγαλύτερη, τα μεγαλύτερα επίγεια σύνορα με ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.300 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αποτελούμε αναπόσπαστο μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τέσσερις ε, βασικές ελευθερίες μας οδηγούν στο να ζούμε αυτές τις ελευθερίες όπως και τα παλαιότερα κράτη-μέλη. Ως προς την έννοια της συνοχής αποτελεί ένα βασικό συστατικό στην επίτευξη αυτού του στόχου και αυτό αφορά και την σύγκληση γενικότερα για να φτάσουμε σε συγκρίσιμο βιωτικό επίπεδο με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη μας επιτυχία. Θα ήθελα εντάχει να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες μας για να κατανοηθεί το όλο θέμα καλύτερα θα μιλήσω στα αγγλικά. Μιλούμε για τέσσερις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας. Έχουμε τέσσερις πυλώνες που αποτελούν το πρόγραμμα της Προεδρίας και αφορά την Ευρώπη που ε, αναπτύσσει, που συνδέει και που αποτελεί μία Ευρώπη της επιρροής μέσα στα πλαίσια της ψηφιοποίησης και στις παγκόσμιες αγορές γνωρίζουμε πολλές προκλήσεις δημοσιονομικές και εργασιακές. Γι' αυτό θα πρέπει να εμβαθυνθεί η ευρωπαϊκή αγορά, η ανάπτυξη, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και η διαβίου μάθηση, καθώς και νέες δεξιότητες που θα πρέπει να ενταχθούν στην ατζέντα της ανταγωνιστικότητας. Η βελτίωση του επίπεδου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερους, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τα περιβαλλοντικά. Γι' αυτό μιλάμε και για την Ευρώπη της ανάπτυξης, τον πρώτο πυλώνα που εντάσσεται στην πολιτική συνοχής και όλα τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Η Κροατική Προεδρία θα υποστηρίξει μια ισορροπημένη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που θα λάβει υπόψη τις ανάγκες όλων των κρατών μελών και περιφερειών. Ένα μέρος, ένα βασικό στοιχείο της Ευρώπης που αναπτύσσει είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Πρόκειται για αρχές που αποτελούν το βασικό μας οδικό χάρτη. Το, ο δεύτερος πυλώνας είναι η Ευρώπη που συνδέει. Υπάρχουν, προϋπάρχουν διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ποιότητα των υποδομών και διαθεσιμότητα μεταφορών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών δικτύων μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση ανταγωνιστικότητας. Για να έχουμε ε, μία οικονομική, κοινωνική και ψηφιακή συνοχή σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τις μεταφορές και τις ε, τηλεπικοινωνίες. Η Κροατική Προεδρία θα ενισχύσει τις πολιτικές υποδομών συνδεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και στον αθλητισμό. Μιλάμε για την Ευρώπη επίσης που προστατεύει. Τρίτος πυλώνας. Θα ασχοληθούμε με την εσωτερική ασφάλεια για πραγματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων με διαλειτουργικότητα των ε, συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για να αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές απειλές και τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Θα θέλαμε να φτάσουμε σε μια συνεκτική λύση για βιώσιμη πολιτική στον τομέα του ασύλου. Γι' αυτό θα προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα πλαίσια της ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης, ε, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Ο τέταρτος πυλώνας είναι η Ευρώπη που επηρεάζει. Θα ενισχύσουμε την ε, πολυπλευρικότητα καθώς και Ε, και θα λάβουμε υπόψη την ατζέντα του ΟΗΕ για την βιωσιμότητα μέσα στα πλαίσια του 2030. Ε, ε, όπως ε, ξέρετε, ασχολούμε με τα θέματα κλιματικών αλλαγών και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι 9,6%. Όταν βλέπουμε την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, που συσσωρεύουν ένα 50% καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Εάν η Ευρώπη λοιπόν έχει φιλόδοξους στόχους έτσι ώστε μέχρι το 2005 να έχουμε ουδετερότητα ως προς τη χρήση άνθρακα και να ε, κόψουμε στο μισό τις εκπομπές μέχρι το 2030 καθώς και τις εκπομπές από την εναέρια κυκλοφορία καταλαβαίνετε ότι ότι αντιμετωπίζουμε ε, άρδιν το πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να αποτελέσουμε η ηγετική δύναμη επηρεάζοντας ε, τα παγκόσμια δρόμενα. Το δεύτερο σημείο που αφορά την Ευρώπη που επηρεάζει είναι η αξιοπιστία της και φυσικά οι διεθνείς ε, σχέσεις έχουν μεγάλη σημασία για μια υπεύθυνη πολιτική γειτονίας, Δυτικά Βαλκάνια, άξονα ανατολίζει Ανατολής Δύσης, Βορρά Νότου. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική ε, διεύρυνσης για ασφάλεια και δικαιοσύνη και καλύτερη συνδεσιμότητα της Ευρώπης. Στο Ζάγκρεπ θα διοργανηθεί μια διάσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια το Μάη όλα αυτά και ελπίζουμε να έχουμε και την υποστήριξή σας για να χαράξουμε έναν οδικό χάρτη για τις χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων ώστε να προσχωρήσουν στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία. Η Ευρώπη λοιπόν που αναπτύσσει, που συνδέει και η Ευρώπη που επηρεάζει οδηγούν σε μια δυνατή Ευρώπη στα πλαίσια των προκλήσεων και έτσι μπορεί να δράσει για την ευημερία των κρατών μελών και των πολιτών. Επιπλέον θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στις προτερότητες της ε, Κροατικής Προεδρίας μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Γενικών Υποθέσεων. Η πολιτική συνοχής, το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, καθώς και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Μέλλον της Ευρώπης. Ε, Αντιπρόεδρος Σουίτσα είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις μας και τις μελλοντικέ μας σχέσεις και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της πολιτικής συνοχής καθώς και την έγκαιρη έγκρισή της με ένα νομοθετικό πακέτο για την περίοδο 21-27. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη ως προς αυτό το θέμα και θα θέλαμε έγκαιρα να έχουμε την έγκριση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα, προ προς το τρίτο τμήμα της παρουσίασής μου στην πολιτική συνοχής και το, τα νομοθετικά σχέδια μέσα στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων, θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς θα είμαστε ένα ειλικρινής μεσολαβητής. Προσπαθήσαμε να, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μία σύγκληση και πιστεύω ότι φέτος, κατά τη διάρκεια μάλλον του εξαμήνου μας, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμφωνίες μέσα στα πλαίσια των δύο συνομοθετικών αρχών, μέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού. Μιλώντας για την ε, πολιτική συνοχής και ως προς το νομοθετικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεχτεί ε, και το ε, ΕΤΠΑ, έχει εγκρίνει μάλλον τις προτάσεις για το ΕΤΠΑ, για το Γεωργικό Ταμείο και το Διασυνοριακό Ταμείο. Πιστεύουμε ότι αυτό ισχύει και με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Έχουν αρχίσει οι εργασίες σήμερα έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια σωστή πλαισίωση. Σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση στην ομάδα εργασίας για τα διαρθρωτικά μέτρα. Επιπλέον, όταν μιλάμε για συνολικές διαπραγματεύσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διατάξεις που έχουν σχέση με τον έγκαιρο προγραμματισμό και την σωστή εφαρμογή των μέτρων. Άρα θα προωθήσουμε τον διαθεσμικό διάλογο με βάση και την πρόοδο που επιτελέστηκε κατά την Φιλανδική Προεδρία. Θεωρούμε ότι οι έγκαιρες αποφάσεις σε όλες τις διαρθρωτικές πολιτικές ε, ότι είναι αναπόσπαστος όρος έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε και το ΠΔΠ 21-27 για να ευεργετηθούν όλα τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Τώρα, να σας μιλήσω για το κάθε χαρτοφυλάκιο χωριστά τον κανονισμό για, το, για το, τις κοινέ διατάξεις, ε, CPR, το ε, Συμβούλιο έχει δεχτεί αυτό το γενικό πλαίσιο έτσι ώστε να υπάρχουν ε, επτά συνδιαχειριζόμενα ταμεία. Η διαχείριση αυτών των ταμείων αφορά ένα νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο για ευελιξία και αναλογικότητα στα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη απλούστευσης και ευελιξίας. Ε, μίλησα για το κροατικό παράδειγμα το 2013 στο ESF. Εμείς είχαμε τον ε, υψηλότερο, το υψηλότερο ποστό ανεργίας, ενώ τώρα έχουμε δίκτυα ανεργίας μόνο 5,7% και 15-16% αφορά τους νέους. Άρα μπορέσαμε να επιλύσουμε το ζήτημα. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Κροατική Προεδρία θα συνεχίσει τον διαθεσμικό διάλογο με βάση την απτή πρόοδο που επιτελέστηκε επί Φινλανδικής Προεδρίας και θα καταλάβουμε κάθε προσπάθεια για να κλείσουμε κεφάλαια υπό την Προεδρία μας. Πριν από ένα μήνα συμφωνήσαμε ότι συμφωνήθηκε μάλλον ότι ε, η εργασία του τεχνικού επίπεδου μπορεί να γίνει και σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον κανονισμό CPR, έτσι ώστε να μπορούν οι χώρες να προβάλλουν τα επιχειρησιακά του σχέδια. Σε σχέση με το ΕΤΠΑ, χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι τα καταφέραμε ως προς το, τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και έτσι τα εντάξαμε σε έναν κανονισμό. Επίσης θα προωθήσουμε το Περιφερειακό Ταμείο και τα διαρθρωτικά με βάση την προσβασιμότητα και την αναλογικότητα. Έχουμε αρχίσει και ε, σε σχέση με το ΕΤΠΑ και τον κανονισμό κοινών διατάξεων και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες ε, προς αυτό το σκοπό. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να ε, πληρώσουμε το κενό που υπάρχει στο ΕΤΠΑ και το Κοινωνικό Ταμείο καθώς και τα διαρθρωτικά σε ό,τι αφορά το κανονισμό Interreg. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ε, καλώς την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την απλοποίηση των διατάξεων και πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εντολή μας σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Interreg, θέλουμε να εξασφαλίσουμε συνέχεια με την προγραμματική περίοδο την υφιστάμενη. Και θέλουμε να συνεχίσουμε τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις βάσει των όσων πέτυχε η Φιλανδική Προεδρία και να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε όσο πιο μεγάλη πρόοδο γίνεται για τι διατάξει που θεωρούνται κρίσιμε για την προγραμματική περίοδο και για την πιο γρήγορη εφαρμογή των προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας. Και τέλος, ο κανονισμός για την διασυνοριακή συνεργασία. Εδώ το Συμβούλιο καλώς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον διασυνοριακό αυτομηχανισμό. Ο κανονισμός μειώνει τις ε, διοικητικές, τα ε, διοικητικά εμπόδια και τα νομικά, τις νομικές αβεβαιότητες. Είναι περίπλοκο το θέμα ασφαλώς και έτσι ζητήθηκε από τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου να εξετάσει περαιτέρω την πρόταση αυτή και αναμένεται απάντηση της γνωμοδότησης μάλλον του, της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου για να εξετάσουμε τις ε, περαιτέρω συνέπειες μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό για τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη από πλευρά των κρατών μελών, διευκρίνηση των, ε, της ευαίσθητης και πίσης ε, των μηχανισμών, θα κρίνουν και τα αποτελέσματα και προσβλέπουμε στη συνεργασία και στη συζήτηση των θεμάτων αυτών. Τέλος. Θα ήθελα να δηλώσω ότι ως Προεδρία εκτιμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι έχει ρόλο σημαντικό να διαδραματίσει. Έχουμε οργανώσει ανεπίσημη συνάντηση στο Ζάγκρεπ στα τέλη Μαρτίου και στην οποία έχουμε προσκαλέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραστεί. Θα είναι μεγάλη μας τιμή να σας υποδεχτούμε στο Ζάγκρεπ και να ακούσουμε και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πολλά θέματα. Κλείνοντας, να τονίσω τη σημασία μιας καλής και επικοδομητικής ε, συνεργασίας, μιας και είμαστε ίσοι ως νομοθέτες. Θεωρώ ότι θα είμαστε εξαιρετικοί εταίροι για να συνεχιστεί αυτή η νομοθετική προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, να ξεκινήσει η συζήτηση, λέει ο πρόεδρο. Να δώσω τον ε, λόγο καταρχά στην κυρία Κρέλ από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερω που ξεκινάτε την πρώτη μα Προεδρία της Κροατίας και που η περιφερειακή πολιτική αποτελεί τόσο σαφή προτεραιότητά σας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για τους στόχους. Η πολιτική συνοχή κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει να είναι έτοιμη από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ωστόσο, έχουμε κάποιες δυσκολίες ακόμα μπροστά μας. Είναι τιμή σα το γεγονός ότι ω Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξη ε, αγωνίζεστε για την περιφερειακή πολιτική, αλλά δυστυχώς ε, η πολιτική της ανάπτυξης ε, θα μπει σε όλο το πακέτο το διαπραγματευτικό για το ΠΔΠ. Τις επόμενες λοιπόν ημέρες ε, θα πρέπει να γίνει μια κατανομή των αρμοδιοτήτων. Από όσο γνωρίζω, το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ θα το διαπραγματευτεί ο κύριος Μισελ ως ε, επικεφαλής του Συμβουλίου και η πολιτική συνοχή είναι στα χέρια της ε, κρατικής προεδρίας. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον έχουν γίνει ήδη συζητήσεις για το πώς φανταζόμαστε ότι θα μορφωθεί η κατάσταση αυτή, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Ο κύριος ε, Ομαζέ, ο πρόεδρος, σας είπε ότι θα ανασταλούν στην παρούσα φάση οι διαπραγματεύσεις μέχρι τέλη Φεβρουαρίου καταρχάς, αλλά αν μέχρι το τέλη Φεβρουαρίου ούτε η Προεδρία του Συμβουλίου, ούτε η Επιτροπή μας έχει ενημερώσει για το πακέτο αυτό, για κάτι διαφορετικό, δηλαδή σε σχέση με αυτά που πρότεινε η Φιλανδική Προεδρία σε, σε ό,τι αφορά και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα ξαναξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Και αυτό προφανώς μας ανησυχεί όλους μας εδώ στην Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το πώς πιστεύετε ότι θα πετύχουμε αποτελέσματα για το ΠΔΠ. Μία πρώτη αντίδραση για την Πράσινη Συμφωνία παρουσιάστηκε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Αυτό τα κράτη-μέλη το υποδέχτηκαν με θετικό τρόπο. Βέβαια, κανείς δεν θέλει να πληρώσει τελικά. Το χέρι στην τσέπη δεν θέλει να βάλει κανείς. Πώς λοιπόν φαντάζεστε ότι θα επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Από το Ρινιού, κύριε Σπιζού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Άκουσα με προσοχή αυτά που μας είπατε για τις τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες της Κροδική προεδρίας και από ό,τι κατάλαβα ότι θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα αναπτυχθεί, που θα ενώνει και θα προστατεύει και η οποία θα ακτινοβολεί. Μια Ευρώπη η οποία θα ενώνει λοιπόν καταρχάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που εργαζόμαστε εδώ για την πολιτική συνοχή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε όμως στις περιφέρειες ότι παντού υπάρχει ευρωσκεπτικισμός και σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά την πολιτική για το κλίμα. Υπάρχει λοιπόν κατεπήγον χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την ανάγκη ανάληψης δράσης για τη συνοχή και για να αποκτήσει αυτό συγκεκριμένη διάσταση και συγκεκριμένα μέτρα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ζητάμε λοιπόν να επιβεβαιώσετε την ε, προθυμία σας να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, γιατί προφανώς ε, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος για όλα τα ταμεία συνοχής. Μιλήσατε για το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, ε, μιλήσατε και για το Interreg, για το ΡΕΚ έχουν τονίσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας για την πολιτική συνοχή, γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο συγκεκριμένα ε, μεταφράζεται, έχει συγκεκριμένη επίπτωση ε, στις ε, περιοχές και στις περιφερειές μας και θα πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε από κοινού λύσεις για τους πολίτες μας και θα ήθελα να σας επενθυμίσω κύριε Υπουργέ ότι είναι κατεπήγον ο χαρακτήρας αυτής της ανάληψης δράσης για όλες τις περιφερειές μας προκειμένου τα μία, τα ευρωπαϊκά, να μπορέσουν όχι μόνο να καταστούν πιο διαφανή, αλλά και πιο προσβάσιμα μέσω της διαδικασίας απλοποίησης τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Από τους Πράσινους, ο κύριος Νίνας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Νίνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε λοιπόν εδώ σήμερα και που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της κρατικής προεδρίας. Αυτό που αναμένουμε από εσάς είναι όχι μόνο να αποτελέσετε καλό εταίρο στις διαπραγματεύσεις, όπως είπαν ε, διάφοροι συνάδελφοι, αλλά θέλουμε να επιδείξετε και μια ηγεσία στα πλαίσια του Συμβουλίου. Η Προεδρία δεν έχει μόνο το καθήκον να αποτελέσει καλό διαπραγματευτή με το Κοινοβούλιο, αλλά και να καθοδηγήσει το Συμβουλίο προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση δε, και αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν από την κρατική κυβέρνηση, είναι υπέρ της συνοχής, υπέρ της ισχυρής Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης. Μιας Ευρώπη που θα έχει τα μέσα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν κατεπηγόντως σας καλώ να μεταφέρετε τις ιδέες σας αυτές προς τα άλλα τα μέλη του Συμβουλίου και να τους πείσετε ότι για να πετύχουμε καλές, καλά αποτελέσματα χρειαζόμαστε χρήματα και σημαίνει αυτό φυσικά και αρμοδιότητες και εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκπληρώσει τα καθήκοντά της. Είμαστε λοιπόν όντως ε, εταίροι στις διαπραγματεύσεις και προφανώς θέλουμε στις διαπραγματεύσεις να υπάρχουν σαφείς ε, στόχοι και θα υπάρξει και πίεση. Προφανώς ε, μας αρέσουν οι προκλήσεις. Αντιλαμβανόμαστε και την ανάγκη για να γίνουν συμβιβασμοί. Αλλά σας παρακαλώ πείτε στο Συμβούλιο τι χρειάζεται για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Να είσαστε καλοί ηγέτες λοιπόν στο Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω επίσης και τον προηγούμενο ομιλητή. Γιατί συμφωνώ, η Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να είναι μόνο μια Ευρώπη με αλληλεγγύη. Και ενωμένοι είμαστε ισχυροί και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα συμβούλιο το οποίο πραγματικά θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ η Φραντσέσκα Ντονάτο για το ID. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να υποβάλω μια συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με ένα από τα θέματα που θα μας προσελκύσουν ιδιαίτερα σε αυτό το εξάμεινο. Γιατί η Κροατία όπως και η Ιταλία είναι μια χώρα της Μεσογείου έχει μια μεγάλη παράκτια γραμμή και πολλά νησιά. Νομίζω ότι ε, τη στιγμή που υπάρχουν και άλλες νησιωτικές περιοχές και χώρες γνωρίζουμε, γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτός ο νησιώτικος χαρακτήρας των χωρών που είναι ένα ειδικό στάτους και αποτελεί στοιχείο κλείδι έτσι ώστε να μπορούν να επέλθουν εξαιρέσεις ως προς τις κρατικές επιδοτήσεις. Πιστεύω ότι η εργασία που θα γίνει στα πλαίσια των πολιτικών συνοχής είναι ύψη της ε, σημασίας, διότι θα πρέπει η πολιτική αυτή να προσδώσει αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς για τις χώρες που έχουν νησιωτικό χαρακτήρα ε, διότι υπάρχει και ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τη στερεά. Ευχαριστώ για, το, για την κούρα, ο κύριος Παπαδημούλης. Καλώς ορίσατε κύριε Παύτη στην ε, Επιτροπή μας εκ μέρους της ε, <clears throat> Κροατικής Προεδρίας. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επί 1,5 χρόνο, σχεδόν δύο χρόνια, από τότε που η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή της για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Συμβούλιο λειτουργεί ως ένα μεγάλο φρένο. Δηλαδή στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε το θέμα, καταθέσαμε τις προτάσεις μας, κάναμε βελτιώσεις στην πρόταση της Κομισιόν. Το Συμβούλιο επί 1,5 χρόνο δεν κατέθεσε καμία πρόταση και στο τέλος η Φιλανδική Προεδρία κατέθεσε μία πρόταση η οποία είναι απογοητευτική και την οποία κανείς δεν υποστηρίζει ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε στην Κομισιόν. Ειδικά δε για τη συνοχή προωθεί περικοπές στις ίδια παράδεκτε περικοπές που κάνει η Κομισιόν. Επομένως, το ερώτημα που σας θέτω είναι εάν έχετε πρόθεση ως Κροατική Προεδρία να πάρετε πρωτοβουλίες στο θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να καταθέσετε μια πρόταση για συμβιβασμό που να είναι πιο κοντά στην πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, ιδιαίτερα στα θέματα της συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής, ή απλώς θα είναι μια προεδρία τράνζιτ, η Κροατική Προεδρία, που δεν θα κάνει τίποτα για αυτό το θέμα και θα το αφήσει στους Γερμανούς. Το ερώτημα είναι απλό έχετε φιλοδοξία αυτό το θέμα να κλείσει επί Κροατικής Προεδρίας. Αν θέλετε να γίνει, που θα είναι πολύ καλό και για την Κροατία και για την Ευρώπη την Ενωμένη, θα πρέπει να καταθέσετε κάτι που να είναι πιο φιλόδοξο και πιο απαιτητικό, που να πλησιάζει προς αυτά που ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι συνομοθέτης. Η εποχή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεχόταν με το πιστόλι στον κρόταφο απαράδεκτες προτάσεις έχει τελειώσει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί τα ωραία λόγια, μια Ευρώπη ισχυρή, ενωμένη που να προστατεύει, αν δεν μετατρέπονται σε πολιτικές και σε δεσμευτικά μέτρα σε ό,τι αφορά τις γραμμές του προϋπολογισμού, μένουν λόγια. Και οι πολίτες θέλουν έργα, όχι λόγια. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ σαφής, πολύ συγκεκριμένος για τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Θα προσπαθήσω να προφέρω αργά το όνομά σας για να μην το κακοποιήσω. Η Αγγέλικα Μποτζανόφσκα. Ευχαριστώ πολύ. Βελτιώθηκε πολύ η προφορά σας κύριε Πρόεδρε από σήμερα το πρωί. Πράγματι είναι μια σημαντική στιγμή αυτή για την Κροατία και θέλω να σας συγχαρώ κύριε Υπουργέ για την ανάληψη της Προεδρίας. Αυτοί οι τέσσερις πυλώνες που μας παρουσιάζετε αποτελούν καλή απάντηση στις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας. Πρέπει να επιταχύνουμε όμως τις διαπραγματεύσεις για να, ξεκινήσουν, ε, να ξεκινήσει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατό. Γίνεται λόγος για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτό θα καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσει για την πολιτική συνοχή και οι διαπραγματεύσει για την πολιτική συνοχή οι καθυστερημένε θα καθυστερήσουν την εφαρμογή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Χρειαζόμαστε τα χρήματα και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, αλλά και τα λοιπά που περιλαμβάνονται στο Ταμείο συνοχή. Οι εθνικοί φάκελοι θα περικοπούν και άρα και άλλοι τομεί και κλάδοι θα υποφέρουν. Ποιο σχέδιο έχετε? για να ελαχιστοποιήσετε τις καθυστερήσεις και τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Και επίσης, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Διαβάζουμε για την κλιματική ουδετερότητα. Και στα συμπεράσματα λέει το Συμβούλιο ότι όλες οι χώρες ξεκινούν η κάθε μία από το δικό της σημείο εκκίνησης και άρα κάθε, κάθε χώρα έχει την ελευθερία να αποφασίσει για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει, για την πορεία που θα ακολουθήσει. Τι θα κάνετε για να σεβαστείτε αυτό το οποίο υπόθηκε το ε, Δεκέμβριο. Επίσης αναφερθήκατε στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια εικόνα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ίσως θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τη συγχρηματοδότηση των έργων και προγραμμάτων στις περιφέρειες οι οποίες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου θα μπορούσαμε ορισμένες ενισχύσεις να τις φτάσουμε στο βέλτιστο και στο ανώτατο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ροβένα Πλούμ παρακαλώ. Πλάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μα κάνατε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Ξέρω ότι ο ρόλος που θα διαδραματίσετε θα είναι κρίσιμος για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί? Διότι Έχετε στα χέρια σας ε, το φάκελο για το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και έχετε στα χέρια σας ε, το φάκελο για την πολιτική συνοχή. Και εγώ έχω θητεύσει σε αρμόδια θέση, ήμουν πρώην υπουργό για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για την ανάπτυξη των περιφερειών και για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μου και όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης και των χωρών μας. Σήμερα, περισσότερο παραποτέ, χρειαζόμαστε την πολιτική συνοχή συνοχής, η οποία είναι κρίσιμη, είναι καθοριστική σημασία, όχι μόνο για τη νέα πράσινη συμφωνία, για το New Green Deal, αλλά και για όλες τις, προτάσεις, όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Λαμβάνοντας υπόψη το εξής γεγονός, Όταν εγώ ήμουν υπουργό στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στη Ρουμανική Προεδρία, η πρώτη διαπραγμάτευση πάντοτε γινόταν με το Κοινοβούλιο. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλέ καθυστερήσει και θα καθυστερήσει κατά πάσα πιθανότητα και η υιοθέτηση και η έγκριση των διαφορών προγραμμάτων. Ερωτώ λοιπόν λαμβάνετε υπόψη σας το ενδεχόμενο προσωρινών μεταβατικών μέτρων για το 2021. Πώς το βλέπετε αυτό, ποια άποψη έχετε υιοθετήσει, πώς θα το χειριστείτε, πώς θα το μεθεδεύσετε αυτό το ζήτημα με τις καθυστερήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τόμισλαβ Σόκολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Χαίρομαι διότι έχω την ευκαιρία να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ιδιότητά σας του εκπροσώπου της Κροατικής Προεδρίας και του εκπροσώπου της Κροατικής Κυβέρνησης, ε, της κυβέρνησης της χώρας που αποτελεί και την ε, πιο πρόσφατη αφιχθήσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι διότι 6,5 χρόνια μετά την προσχώρηση της χώρας σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κροάτες έχουν την ευκαιρία να προεδρεύσουν, να αναλάβουν την εκπεριτροπή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με τις προτεραιότητές σας, πράγματι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι και το απόλυτο σημείο προτεραιότητάς μας και συμφωνώ με την τοποθέτησή σας για την πολιτική συνοχή η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πιστεύω ότι θα μπορέσετε να βρείτε τη σωστή λύση ε, ε, στα διάφορα θέματα. Ξέρετε, στη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενίοτε συζητούμε τις διάφορες πτυχές της ε, πολιτική συνοχή και ενίοτε συζητούμε και την εφαρμογή ή την υλοποίηση, η οποία ήταν αρκετά προβληματική σε κάποιε χώρε. Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ω επιχείρημα για να μειωθεί ο χρόνο το περιθώριο, το χρονικό ή οι πόροι που δίδονται κάθε φορά για να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής. Έχω θητεύσει έχετε θητεύσει ως Υπουργός ε, και στο παρελθόν, είστε αρμόδιος και είχατε σχετικά χαρτοφυλάκια. Τι κάνει η κροατική κυβέρνηση για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται, αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Κροατία και ποια είναι τα μελλοντικά βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει όλο αυτό το θέμα της υλοποίησης. Τα τελευταία τρία χρόνια της αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Κροατία ήταν τρία χρόνια τα οποία μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά success story, ιστορία επιτυχίας και μπορούν να εμπνεύσουν και τις λοιπές χώρες για να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης, ε, χρησιμοποίησης, αξιοποίησης και εφαρμογή. Έτσι ώστε να φανούν τα ωφέλη της πολιτικής συνοχής, μια πολιτική η οποία ενσαρκώνει την ε, βασική θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης πάνω στην οποία δράζεται το οικονοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Ο κύριος Πεκάρινεν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχάς για την ανάληψη της ε, Κροατικής Προεδρίας. Ξέρω ότι η διαδρομή σας είναι πολύ σημαντική. Ξέρω ότι έχετε σημαντικές ευθύνες στο Συμβούλιο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας δίνω συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι είστε σε θέση να μας φέρετε καλά αποτελέσματα. Όμως, αν κάνουμε την ανάστροφη πορεία και αν δούμε τι έχει συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανατρέχοντας την περασμένη δεκαετία και στα τελευταία δέκα χρόνια, εύλογο είναι το ερώτημα που τίθεται. Τι γίνεται με την πολιτική συνοχή. Υποτίθεται ότι έχουμε πολιτική συνοχή για να μειωθούν οι διαφορές. Να μειωθούν οι διαφορές π.χ. σε επίπεδο ΑΕΠ μεταξύ των διαφορών χωρών και των διαφορών περιφερειών και περιοχών. Αν κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή και δούμε τα, τα στοιχεία, συνειδητοποιούμε ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών σήμερα είναι όντως μικρότερες από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Και πρώτα απ' όλα οι διαφορές μεταξύ των μεγάλων πόλεων στις χώρες που εντάσσονται στο Ταμείο Συνοχής έχουν καταφέρει οι χώρες αυτές ε, στις μεγάλες τους πόλεις ε, τα, οι επιδόσεις να είναι φάμιλες με ε, τις μεγάλες πόλεις των ε, δυτικών παλαιών χωρών που είχαν πολύ υψηλές επιδόσεις ούτως ή άλλως και ψηλά αποτελέσματα. Όμως οι περιφέρειες υστερούν. Δηλαδή έχουμε πετύχει συνοχή γενικά σε επίπεδο πληθυσμού, έχουμε πετύχει συνοχή σε επίπεδο πόλεων, αλλά δεν έχουμε πετύχει συνοχή σε επίπεδο περιφερειών. Ποιες είναι οι διαδικασίες που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειώσετε τις διαφορές αυτές και ε, όχι μόνο μεταξύ των βασικών και μεγάλων πόλεων αλλά και των ε, περιοχών της Υπέθρου ή των κομμοπόλεων και μικρότερων κοινοτήτων. Γιατί εκεί στην Υπέθρο και στις κομόπολεις και στις ε, μικρές περιφέρειες παραμένουν μεγάλες διαφορές και η πολιτική συνοχή δεν έχει πετύχει. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Άλβαρο Αμάρο, επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας κατά την Κροατική Προεδρία. Άκουσα με προσοχή τους ε, τέσσερις πυλώνες που κατονομάσατε, Ευρώπη που αναπτύσσει, επηρεάζει, συνδέει, αλλά σήμερα το πρωί είχαμε μία συζήτηση με την Επίτροπο και είπαμε πολύ, αναφέραμε πολύ το εξής. από αυτά που άκουσα από την Επίτροπο σήμερα το πρωί φαίνεται ότι είμαστε αλληλέγγυοι από πλευράς Επιτροπής και Κοινοβουλίου για να υπάρξει μία ουσιαστική πολιτική συνοχής. Αλλά μιλήσαμε για fresh money, γιατί, για νέο χρήμα, διότι αν δεν υπάρξει νέο χρήμα, τότε ε, αλληλοαπατώμεθα. Πιστεύω ότι η Κροατία, και επειδή ακούσαμε τις προτεραιότητές σας, πιστεύω ότι η Κροατία ε, τάσεται υπέρ της συνοχής. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για το εξής. μην παραμένετε στα λόγια για νέο χρήμα ως προς νέες πολιτικές, διότι υπάρχουν νέες αξίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και δεν νομίζω ότι μπορούν να περάσουν σε δεύτερη μοίρα πολιτικές που έχουν ακόμα πάρα πολλά να δώσουν για αυτή την Ευρώπη που αναπτύσσεται, όπως λέει και ο πρώτος σας πυλώνας, μια Ευρώπη που αναπτύσσεται, μια πιο δίκαιη Ευρώπη. Και συνεπώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη περιφέρειες που είναι λιγότερο αναπτυγμένες, ακόμα και σε πλούσιες χώρες Αυτές οι φωνές ακούγονται όλο ένα και περισσότερο. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν γίνουν περικοπές στο Ταμείο Συνοχής. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβιβάσετε στο Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να γίνουν περικοπές στα διαρθρωτικά ταμεία. Γιατί ε, δεν μπορούμε παρά να θέτουμε σε ίση μοίρα όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Φρανσουά Αλφονσίν. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην κρατική Προεδρία που αναλαμβάνει αυτή την Προεδρία σε ένα κρίσιμο, ε, ένα κρίσιμο χρονικό, σε μια κρίσιμη, κρίσιμη χρονική στιγμή για τις ευρωπαϊκές πολιτικές που τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να μας οδηγήσουν προς στόχους μεγάλης εμβέλειας και φέρετε μεγάλη ευθύνη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα που με απασχολεί ιδιαίτερα γιατί προέρχομαι από την ε, Κορσική που έχει επίσης νησιωτικό χαρακτήρα. Είπατε, μιλήσατε για προτεραιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα, αλλά πολλές φορές θεωρήσαμε ότι τα νησιά ε, βρίσκονται πέραν της ανάπτυξης. Και αυτό είναι αντικειμενικό, γιατί τα νησιά πλήττονται από θέματα σύνδεσης και συνδεσιμότητας και μαζί με τον κύριο Πίτσουλα, τον συμπατριώτη σας, έχουμε προβεί στη σύσταση μιας ομάδας που ονομάζεται Σίλικα και έχουμε σκοπό κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου να ε, οργανώσουμε μία διάσκεψη για ε, το θέμα αυτό των νησιών θα μπορούσε να παρέμβει η Κροατική Προεδρία έτσι ώστε να υπάρξει μία απήχηση του ζητήματος αυτού. για να ληφθούν υπόψη τα αιτήματά μας ως προς το μέλλον της ε, Ευρώπης της Συνοχής. Ευχαριστούμε πολύ Φρανσουά. Πολλές παρεμβάσεις ακούσατε, αλλά όλες συγκλίνουν προς το ίδιο αίτημα και επιθυμία που θα μπορούσα να συνοψίσω ως εξής. Ε, δεν περιμένουμε πολύ περισσότερα από αυτά που μπορείτε να κάνετε. Δηλαδή δεν περιμένουμε μία ουδέτερη προεδρία, αλλά μία προεδρία η οποία δεσμεύεται ενώπιον του Συμβουλίου υπέρ της συνοχής. Έγιναν πολλές διαθεσμικές συναντήσεις και χαίρομαι γιατί δώσατε συνέχεια σε όλα αυτά τα θέματα υπό την Προεδρία σας ε, τα καταφέραμε να προωθήσουμε τον, το ΣΕΠΕΡ και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Σε αυτή τη στιγμή ζωτικής σημασίας πιστεύω ότι υπάρχει θέληση σύγκληση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κροατική Προεδρία για να δημιουργηθούν οι βέλτιστοι δυνατοί όροι έτσι ώστε αυτή τη δύσκολη στιγμή να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον κανονισμό αυτό. Πιστεύω ότι το ΣΕΦΠ οπωσδήποτε θα προωθηθεί μέσα στα πλαίσια του αρμόδιου επιτρόπου και χαρτοφυλακίου. Θα θέλαμε όμως και εσείς να δράσετε κατά τον βέλτιστο δυνατό, δυνατό τρόπο έτσι ώστε να επανέλθουμε σε μία δυναμική πορεία, έτσι ώστε να προωθήσουμε τις ε, πολιτικές μας εκεί που φαίνεται ότι καρκινοβατούν. Μέσα στα πλαίσια του ε, προϋπολογισμού και του κανονισμού που χρήζει βελτίωσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές και τους συζητητές ε, για τις ερωτήσεις που έθεσαν. Να πω δύο λόγια για το ΠΔΠ γενικά. Καταρχάς, αντιλαμβανόμαστε ότι η Φιλανδική Προεδρία το Δεκέμβριο παρουσίασε το πακέτο των διαπραγματεύσεων, αυτό το κοιτίο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις ε, του Δεκεμβρίου έγινε έκκληση από το Συμβούλιο να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να πετύχουμε τελικές συμφωνίες. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Μισελ και το γραφείο του ξεκίνησαν τις διμερείς ε, συναντήσεις ε, και η κρατική αντιπροσωπεία συμμετείχε σήμερα το πρωί στις διαπραγματεύσεις αυτές, άρα οι διμερείς ε, διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ξεκινήσει. Είναι φιλόδοξες και θα ήθελα να τονίσω προς όλους τους βουλευτές που έκαναν σχόλια για το χρονοδιάγραμμα, για την κυρία Κρέλ αλλά και για όλους, ότι είμαστε φιλόδοξοι. Αλλά με την απόφαση του Συμβουλίου που ελεύθεσε το Δεκέμβριο, πλέον ο πρόεδρος ε, Ζαν Μισελ έχει την ε, αρμοδιότητα να υποβάλει και να ξεκινήσει τις, να κάνει προτάσεις. ο πρόεδρο του Συμβουλίου, ο κ. Πλένκοβιτ, θα διατυπώσει τι απόψεις του στα πλαίσια του Συμβουλίου, αλλά από πλευρά της Προεδρίας θα ήθελα να παρουσιάσω το έργο της Προεδρία και τις προτεραιότητε, της δικές μας. Όπω είπατε, η Κροατία είναι γνωστό τι απόψεις έχει και πώ το αποφατείται σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της συνοχής και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Χρειαζόμαστε επίσης τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό ως Προεδρία λοιπόν καλούμε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην ε, συνάντηση στα τέλη Μαρτίου στο Ζάγκρεπ και επίσης ε, Γίνεται διάλογος σε όλα τα επίπεδα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπιζού και τα σχόλιά του. Να σχολιάσω ότι μπορούμε να προβούμε σε απλοποίηση του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ σε, τομεακές, σε τομεακούς κανονισμούς και εκ παραλλήλου μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το πει. Προς τον κύριο Νίνας. Διευκρίνησε ότι χρειάζονται ηγεσία τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου. Εμείς ως Προεδρία καταβάλουμε προσπάθειες. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, αλλά την ε, αρμοδιότητα ανάληψη πρωτοβουλίων για το θέμα του ΠΙΔΛΤΑΠΗ την έχει ο κύριος Μισελ, η κυρία Ντανάτο και ο κύριος Αμφόντση. Μίλησαν για τα νησιά. Η κρατία όπω γνωρίζετε, είναι μια χώρα με πάνω από χίλια νησιά. 50 και πλέον κατοικούνται. Διευκρινίσαμε στο Συμβούλιο λοιπόν ποια είναι η τοποθέτησή μας σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Αυτό αποτυπώνει λοιπόν τις ιδιαίτερότητε των νησιωτικών περιοχών. Θα ληφθούν λοιπόν υπόψη ε, ε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτά για να αποφευχθούν οι διακριτικέ μεταχειρήσεις και όπως υπάρχει η περιφερειακή στρατηγική για τα νησιά, θα έχουμε και πρωτοβουλίες για τα ευφύ νησιά Είδαμε κάποια καλά παραδείγματα από τα Ιταλικά νησιά και την Κορσική επίσης την επισκεφθήκαμε προσφάτως στα νησιά Όκνη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όταν μιλάμε παρεπιπτόντως για τον Brexit, να πούμε ότι η νήσι Όκνη στο Ηνωμένο Βασίλειο δέχονται επενδύσεις από τρεις διαφορετικούς οικονομικούς φακέλους, τις οποίες και αξιοποιούν είναι η περιφέρεια με τις, ε, πιο πολλά, τα πιο ψηλά ποσοστά υπέρ του Remain, υπέρ της ε, παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, λοιπόν. Ένα, ενεργειακό, ένα κέντρο ναυτιλιακό συστάθηκε. Προωθούνται τα ηλεκτρικά οχήματα επίσης στα νησιά και πρωτοβουλίες για τις μπαταρίες, όπως επίσης και φέρει για με ενέργεια. Ένα από τα ερωτήματα του κ. Αλφόνση ήταν το θέμα της συνδεσιμότητας. Είπατε ότι εργάζεστε με τον κύριο Πιτσούλα για τη διάσκεψη. Είμαι βέβαιο ότι στα πλαίσια τη Προεδρία θα υποστηρίξουμε τέτοιε διασκέψει και για μα ε, τα νησιά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και για την Κροατία χώρα αλλά και για την Προεδρία. για, προς την κυρία Πλάμ, η οποία υπογράμμισε το μέλλον της Ευρώπης και ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προχωρήσουμε. Και ζητούμε βοήθεια και κάνουμε διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζουμε ότι τα κονδύλια θα διδεθούν εγκαίρως σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Βασική φάση των διαπραγματεύσεων είναι η φάση των διαπραγματεύσεων με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι βασικοί φορείς, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Και θα πρέπει τα θέματα αυτά να θα συζητήσουμε και να διαβουλευτούμε σχετικά με τους πολίτες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα αντιευρωπαϊκά λαϊκιστικά κίνηματα που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σχόλια του κυρίου Σόκολ τώρα για την εφαρμογή στην Κροατία και τις εμπειρίες μας και τι μπορούμε να πούμε βάσει της εμπειρίας μας, να πούμε ότι είναι ο πρώτος ε, χρηματοοικονομικός αυτός φάκελος και ξεκινάμε με 9% πόρους ανάθεσης και τώρα είμαστε στο 23,4%. Έχουμε καταβάλει ένα τρίτο, τρία δις ευρώ, λοιπόν, ε, ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε το πλήρη φάκελο για τις συμβάσεις στο 100%. Ποιες είναι οι νέες ιδέες τώρα σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της ε, σύνδεσης μεταξύ ERDF και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου ΕΤΠΑ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση. Το ένα ταμείο χρησιμοποιείται για να αναπτυχθούν προγράμματα και το άλλο για να υπάρξουν υποδομές. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη σύνδεση το πρόγραμμα για παράδειγμα WIST στην Κροατία όπου επενδυθήκαν 150 εκατομμύρια ευρώ για να απασχοληθούν πάνω από 6.000 γυναίκες στην Ήπετρο και επίσης ε, δημιουργήθηκαν πολλά κέντρα για την παροχή βοήθειας σε τέτοιες ε, περιθωριοποιημένες ομάδες αυτή η σύνδεση, αυτός ο, η διασύνδεση θα αποτυπωθεί και στην διάρθρωση των προγράμματων αυτών στο μέλλον, ιδιαίτερα στην Κροατία. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Πεκαρίνεν τώρα, για τις διαφορές που υπάρχουν ε, μεταξύ της συνοχής. Ε, αυτό το είδαμε στην Κροατία Σλοβενία, Βαρνία και ΣΡΙΕΜ και πέντε ακόμα ανατολικές επαρχίες εντοπίστηκαν που είναι στο 32-33% επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για σκοπούς ε, σύγκρισης το Ζαγκρέπ είναι στο 108%. Υπάρχουν ε, λοιπόν προβλήματα, αρκετά μεγάλα προβλήματα και αποκλήσεις εντός της Κροατίας και η κυβέρνηση δημιούργησε αυτό το πρόγραμμα Σλοβενία Σινέμα και αμα, αναθέσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ στο έργο αυτό. Και κυρίως ε, αυτές τις περιοχές ε, στοχεύσαμε, τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές και την άμακτη Ζάβρα. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν πιο πολύ τη σημασία των περιοχών αυτών. Γιατί οι πιο πολλοί κάτοικοι της χώρας μας είναι από τέτοιες περιοχές και πραγματικά μας συνεχάρισε η Επιτροπή, μιας και προερεύει του έργου αυτού. Είναι λοιπόν αυτό ένα από τα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση και αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση. Θα το προωθήσουμε και ως ε, βέλτιστη πρακτική στο μελλοντικό οικονομικό φάκελο. Και αυτό επίσης θα αποτυπωθεί στη μελλοντική διάρθρωση των προγραμμάτων. Όπως είπε ο κύριος Μάρς, επίσης υποστηρίζει τους πυλώνες και την αλληλεγγύη ως προς το σκέλος της ηγεσίας και πώς μπορούμε να βρούμε πιο πολλές επενδύσεις στην Κροατία τονίζουμε την περιφερειακή συνεργασία για να γεφυρώσουμε τις διαφορές που υφίστανται. Κλείνοντας το γύρο των ερωτήσεων αυτών, θα ήθελα να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι για το επόμενο διαπραγματευτικό κουτί αρμοδιότητα για ανάληψη πρωτοβουλειών έχει ο κύριος Μισελ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Η Κροατία, ωστόσο, είναι πολύ φιλόδοξη και σκοπεύουμε να κινηθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε και να προωθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται τα, θέματα συνοχής στο όλο πλαίσιο του ΠΔΠ. Με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Μάρκο Πάβιτς. Κύριε Υπουργέ, σας διαβεβαιώ ότι θα έχετε τη στήριξη της Επιτροπής μας και κατά πάσα πιθανότητα και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το στόχο της συνοχής και για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού προϋπολογισμού για τα θέματα που μας απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε θερμότατα το πολύ θετικό νέο που μας έχετε αναγγείλει, τη διοργάνωση άτυπου συμβουλίου για θέματα συνοχής. Δεν απασχόλησε αυτό το ενδεχόμενο τη Φιλανδική Προεδρία. Εσείς το έχετε αναλάβει. Ε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα προχωρήσουμε πλάι-πλάι. Ε, σας εύχομαι καλή προόδο, καλή συνέχεια στην Προεδρία σας και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ, για την ανταλλαγή απόψεων. Bien. Καλώς. Καλώς. Συνεχίζουμε. Je remercie aux uns et ε, Σε παρακαλώ αποχωρήστε από την αίθουσα ησύχως. Όσοι δεν θα παραμείνετε για τη συνέχεια της συνεδρίασης. Yeah. Comment on dit en anglais pour vous quitter la salle Could you leave the room Yes, we left. Could you leave the room in silence, please? Παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως, το λέω και στα αγγλικά. Bien. Très bien. Ils sont partis, mais les Αυτοί έφυγαν, αλλά οι καλύτεροι έμειναν. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τώρα τον κύριο Ενρίκο Ρώση, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της, διά... της ε, περιφέρειας της Τοσκάνης στην Ιταλία, άρα είναι ο περιφερειάρχης της ε, Τοσκάνης και είναι αντιπρόεδρος της διάσκεψης των παράκτιων ε, περιφερειών της Ευρώπης. Η CPMR είναι ένας εταίρος πολύ σημαντικός, ένας συνεργάτης βασικός για τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή από τη στιγμή που ο κοινός μας στόχος είναι, είναι η υπεράσπιση και η διάδοση της περιφερειακής πολιτικής. Πορευόμαστε μαζί με τις CPMR, ε, όλα αυτά τα χρόνια από τότε που πρώτο επινοήθηκε ο όρος πολιτικής συνοχής και νομίζω μάλιστα ότι η διάσκεψη των, περιφερειών, των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης δημιουργήθηκε πριν από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λέω αυτό για να αναδείξω ε, το βάθος το, της εμπειρογνωμοσύνης της διάσκεψης αυτής. Έχουμε πολλά να μάθουμε, έχουμε μάθει πολλά από τη διάσκεψη των παράκτιων περιφερειών. Ουσιαστικά μιλούμε για τη διάσκεψη των παράκτιων και θαλάσσιων περιφερειών της Ευρώπης. Και παρόλο που το έχουμε πει πολλές φορές, χρειάζεται πάντοτε να, να το πούμε ακόμα μια φορά ή να το λέμε και να το ξαναλέμε. Οι θαλάσσιες περιοχές, οι παράκτιες περιφερειέ είναι εξαιρετικά σημαντικές, κυρίως σήμερα περισσότερο παραποτέ με βάση τους νέους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι το πιο αποκομμένο μέρος του κόσμου. Τι εννοώ αποκομμένο, εννοώ κατακαιρματισμένο. Έχουμε δαντελωτές δηλαδή ακτέ, έχουμε πρόσωψη στη θάλασσα, στην Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή γεωγραφική επικράτεια περισσότερη, μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη από ό,τι ε, στις υπόλοιπες χώρες. Ε, όλες αυτές οι περιοχές έχουν τεράστια σημασία και για τη γαλάζια οικονομία και για όλους τους στόχους μας. Η νησιωτικότητα είναι ένα του, είναι πλεονέκτημα. Το να έχει κανείς, το να έχει μια χώρα θαλάσσιες, παραθαλάσσιες και παράκτιες περιοχές είναι πλεονέκτημα, αλλά είναι και πρόκληση. Γιατί οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, κυρίως ως προς την ψηφιοποίησή τους και την πρόσβασή τους στη ψηφιακή εποχή μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων. Όταν ήρθε η Επίτροπος κυρία Φερέιρα στην Επιτροπή μας για να γίνει η ακρόασή της, μας είπε ότι η βούλησή της είναι να δουλέψει για μια Ευρώπη και για μια περιφερειακή πολιτική à la carte. Δηλαδή ε, πρέπει να ε, ε, ράψουμε το κουστούμι που ταιριάζει σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, είτε είναι παράκτια είτε είναι νησιωτική, αναλόγως με το κατά πόσο είναι υπηρετική και ούτω καθεξής. και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έξι είναι οι υποεπιτροπές της διάσκεψης των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης για τη Μαύρη Θάλασσα, για τα Βαλκάνια, για τη Βαλτική θάλασσα, για τον Ατλαντικό, για τα νησιά και ούτω καθεξής. Ε, ε, έχουμε το μεγαλύτερο ε, νησιωτικό λεκανοπέδιο εμείς στην Ευρώπη, αν θέλετε. Το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα στο σύνολο των χωρών. Επομένως, με πολύ μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε, κύριε Αντιπρόεδρε της CPMR, κύριε Ενρίκο Ρώση, Θέλω να διευκρινίσω ότι συνοδεύεστε από τη φίλη μας, την κυρία Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέα της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης, την οποία και καλωσορίζω επίσης. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Γεια σας, σας καλησπερίζω όλους, τον Πρόεδρο και την Επιτροπή σας εξ της διάσκεψης των παρακτήων περιφερειών της Ευρώπης. Από το 1973 υπάρχει αυτή η οργάνωση και εκπροσωπεί 150 περιφέρειες ε, σε γύρω 25 χώρες. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη φωνή των περιφερειών στην Ευρώπη και να προωθήσουμε μία εδαφική πολιτική εντός Ευρώπης. Όπως ακούσαμε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνέλθει σύντομα για να μιλήσει για το ΠΔΠ. Ε, ως CPMR ε, ανησυχούμε για δύο λόγους, διότι έχει περισταλεί ο προϋπολογισμός σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Και στη συνέχεια είδαμε και τη στάση της ε, Φινλανδικής Προεδρίας. Άρα μειώνονται οι πόροι σε πολλά κράτη-μέλη ε, ως προς τον ε, τελικό προϋπολογισμό και χρηματοδότηση. Όπως βλέπετε από αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε ότι υπάρχουν δύο χώρες, η Ελλάδα και η Ιταλία και βλέπουμε πώς φτάσαμε σε μία χαμηλότερη ε, κατηγοριοποίηση. Ε, ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε μία καλύτερη χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια του πι δελτα πι. Θα πρέπει Επίσης, να λάβουμε υπόψη και μία φιλόδοξη χρηματοδότηση για τη συνοχή με βάση τις ε, πρόσφατες προτάσεις. Η πολιτική της συνοχής είναι το κυριότερο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να φτάσουμε στο πράσινο σύμφωνο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση, γι' αυτό όλες οι περικοπές έρχονται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες μας, τις εν γέννη φιλοδοξίες. Το δεύτερο θέμα ανησυχίας αφορά την πολιετή χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου διατρέχουμε τον κίνδυνο το πρόγραμμά μας που αρχίζει την 1η Πρώτου 21 να ε, ενέχει κανονισμούς που δεν έχουν εγκριθεί και αυτό θα είχε αλυσίδωτες αντιδράσεις και αδυνατότητα δαπάνης. για τις περιφερειακές οικονομίες και αυτό αφορά τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολλές ε, δαφικές οντότητες υπάρχουν ε, διαρθρωτικές δυσχέρειες που οδηγούν σε πολλαπλές δυσκολίες και γι' αυτό υπάρχει ε, θέμα και σχέση με ΑΕΠ συγκεκριμένων περιφερειών. Γι' αυτό ακριβώς οι παράκτιες περιφέρειες της Ευρώπης ζητάν τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ε, υποστηρίζουμε μέτρα τα οποία θα μας ε, ε, επιτρέψουν να δαπανίσουμε από την, από την πρώτη μέρα, να έχουμε σχέδια κατεπίγουσας ανάγκης και να υπάρχει προγραμματισμός ακόμα και εάν υπάρχουν καθυστερήσεις έγκρισης του προϋπολογισμού. Υπενθυμίζω τον κρίσιμο ρόλο της ε, πολιτικής συνοχής. Το CPMR δέχτηκε την ε, εδαφική συνδεσιμότητα που προσέδωσε το νέο μέσο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα ταμεία στην πολιτική συνοχής. Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ε, συνεχή συμμετοχή στον προγραμματισμό στις ίδιες τις περιφέρειες και ιδιαίτερα για τις δαπάνες αυτών των πόρων ε, μέσα στα πλαίσια της εδαφικής παρέμβασης. Επίσης, οι κεντρικές κυβερνήσεις θα έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν για τους τομείς που θα λάβουν αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να μην υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις ε, κατά συγκεκριμένων περιφερειών και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να παρέμβει για να ενισχυθούν αυτά τα κονδύλια. Επίσης, ως προς το ε, Ταμείο ε, αυτό της δίκαιης μετάβασης, εδώ μιλάμε για νέο χρήμα της τάξης του 7,5 δις μέσα στα πλαίσια του ιδίου προϋπολογισμού που δεν θα είναι επιπρόσθετα κονδύλια. Δηλαδή ε, έτσι ακριβώς αφαιρούνται κονδύλια από τις διαρθρωτικές πολιτικές. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό και η εισαγωγή ενός νέου ε, ταμείου δεν σημαίνει ότι μειώνονται οι συνολικοί πόροι της γενικότερης χρηματοδότησης. Εδώ δεν μιλάμε για πολιτικές που ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Θεωρώ ότι το Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης θα πρέπει να βοηθήσει την δημιουργία τέτοιων υποδομών ε, και αυτό αφορά και τον κανονισμό μετά το 2020. Ε, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έθεσε τον όρο της μακροοικονομικής ερεσιμότητας. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να παλινοδίσουμε. Δηλαδή, γιατί να μην μπορούν οι περιφέρειες να λαμβάνουν αποφάσεις. Δυστυχώς συνεχώς θίγονται και ευεργετούμενοι, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη στον ε, κεντρικό προγραμματισμό και κρατικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε μία πολιτική συνοχής ως βασικό πυλώνα οικονομικής διακυβέρνησης για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και αυτό αφορά και την περιφερειακή συγχρηματοδότηση που βρίσκεται εκτός συμφώνου σταθερότητας, έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία και να εξασφαλιστούν περισσότερες επενδύσεις. Ως περιφερειάρχης της ε, Τοσκάνης δεν μπορώ παρά να μιλήσω για τις τοπικές ιδιαιτερότητες οι συνθήκες ορίζουν τις ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες, τον ισιωτικό χαρακτήρα πολλών περιφερειών και ούτω καθεξής. Πολλές φορές υπάρχει και απερίμωση περιφερειών ανάλογα με τις γεωγραφικές συνθήκες και την διαθεσιμότητα υπηρεσιών. Και Επιπροσθέτως υπάρχει έλλειψη επενδύσεων. Γνωρίζω ότι ο κύριος Πασολίνο στην έκθεση του μίλησε για τους κανονισμούς μετά το 2020 σε αυτούς τους τομείς. Θα ήθελα αυτό το θέμα να επιβεβαιωθεί από όλους εσάς για να μπορείτε να μας υποστηρίξετε περαιτέρω στη μάχη που δίνουμε για να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε διάφορα στοιχεία και διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν και το θέμα της ρεσιμότητας, ε, της μακροοικονομικής ρεσιμότητας, τη θέση επίσης ε, του Κοινοβουλίου, τη γνωρίζετε, δεν είναι θέση δογματική και ιδεολογική. Όχι, αποκλειστικά δηλαδή. Είναι μια τοποθέτηση που αποσκοπεί σε μια σωστή και δίκαιη προσέγγιση. Γιατί οι επικεφαλείς των περιφερειών, οι περιφερειάρχες μας α, λένε διαρκώς πόσο άδικο είναι το γεγονό ότι δημιουργούνται οι περιφέρειε για το γεγονό ότι δεν σέβονται την δημοσιονομική πειθαρχία τα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν μια διαφορετική συζήτηση αυτή. Αλλά να είστε βέβαιο ότι από πλευρά ε, Κοινοβουλίου και τη επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, έχουμε μία εντολή πλήρη για να προασπιστούμε την ψήφο της Ολομέλειας που απορρίπτει τη μακροοικονομική αρισμότητα. Θα είμαστε λοιπόν σταθεροί και αμετακίνητοι στις διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις προκειμένου να μην υπάρξει τέτοια ρεσιμότητα, να μην αποτυπωθεί αυτή η ρεσιμότητα στον κανονισμό. από την ε, ΣΥΠΙΡΑ με η κυρία Μαριανού. Θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο, όχι μόνο για το θέμα της ρεσιμότητας που αποφασίσετε πραγματικά ότι δεν βολεύει ουσιαστικά, δεν έχει να κάνει με την πολιτική συνοχή στην ουσία της, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έχει πετύχει η Επιτροπή ε, στις... Ε, διαπραγματεύσει τη ω συνομοθέτη. Είμαστε αμετακίνητοι σε ό,τι αφορά την αρχή εταιρική σχέση. Και ξαφνικά το Συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτή η αρχή με τις περιφερειακές αρχές για τη συνεργασία με τι περιφερειακές αρχέ δεν είναι υποχρεωτική. Θα επαφείται στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν κατά πόσον θα συμμετέχουν ή όχι οι περιφερειές. Θεωρώ όμω ότι εφόσον Λέμε εδώ, στο Κοινοβούλιο και πέρα από το Κοινοβούλιο, ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτε θα παρακολουθούν και θα καταλαβαίνουν τι κάνουμε και πώ το κάνουμε και πώ ε, εφαρμόζονται συγκεκριμένα οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Έμα ε, είναι απαραίτητο να είναι στο επίκεντρο τη διαδικασία τη πολιτική συνοχή οι περιφέρειε και να συμμετέχουν εγκαίρω στι συζητήσει αυτέ και στην κατάρτιση και τη χάραξη πολιτική. Το γεγονό λοιπόν ότι σε τελική ανάλυση στο τέλος της διαπραγμάτευσης εξασφαλίζεται ότι η συμμετοχή και η των περιφερειών θα είναι απαραίτητη, είναι σημαντικό βήμα. Και αυτό θα έχει συνέπειες, θεωρώ, και για το πώς αγγίζουμε τους πολίτες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο ήθελα να τονίσω. Το θέμα της περιφερειακής ε, Συνεργασία στο Interreg. Και πάλι, σε ό,τι αφορά το τι κάνει το Interreg, πολλοί βουλευτέ ε, που συμμετείχαν στη συζήτηση με την Επιτροπό υποστήριξαν το Interreg, γιατί το Interreg ενώνει τους ανθρώπους και ελπίζω να μην συγχυστεί η Νόκια που χρησιμοποιώ το σλόγγαν τη. Ε. Αλλά πραγματικά όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αυτοί που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα μετά το τέλος του μήνα ή όποτε συμβεί το Brexit, το ίντερεκ λοιπόν είναι σημαντικό. Και ένα από τα στοιχεία τα οποία υποστρέφτηκαν από το Κοινοβούλιο είναι το εξή. Η ναυτιλιακή συνεργασία αποτελεί έναν τρόπο Συνεργασία και στον διασυνοριακό κλάδο, γιατί είχε αφαιρεθεί αυτό. Όταν λοιπόν ήρθε η πρόταση, ξαφνικά δεν περιλαμβανόταν η θαλάσσια αυτή η συνεργασία. Το συζητήσαμε λοιπόν με το Κοινοβούλιο και ο κ. αποφάσισε ότι αυτό δεν ήταν σωστό τρόπο αντιμετώπιση και διορθώθηκε. Είδατε λοιπόν το χάρτη που είχε προβάλει ο πρόεδρο στι οθόνε. Στόχο μα λοιπόν είναι να βρούμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρακτικά δεν λειτουργούν στι ε, περιφερειε, να κάνουμε αναλύσει και μελέτε να σα διαθέσουμε, να διαθέσουμε για να τι έχετε. Το κάναμε αυτό και για την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό σε όλους τους τομείς που είναι σημαντικοί για το Κοινοβουλίο. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ βασικό δεν είναι συμφωνία πι αλλά είναι σημαντική η συμφωνία γιατί επηρεάζει την ε, στάση μας. Είναι η θεματική, περιφερειακή θεματική επικεντρώση. Η πρόταση είναι να γίνεται σε εθνικό και όχι περιφερειακό επίπεδο η επικεντρώση. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ξεχνούμε εντελώς την αρχή της περιφερειακής προσέγγισης. Και εδώ λοιπόν πάλι. Θα πρέπει όλα αυτά να μπουν στο επίκεντρο των προσπαθειών μα ω συνομοθέτε. Επιστώ λοιπόν την προσοχή σα και σε αυτό. Τέλο, αναφέρθηκε σε διάφορε περιπτώσει και η Επιτροπός το ανέφερε προηγουμένω. Ε, το θέμα των νησιών. Δεν είμαι βέβαιη ότι λάβαμε απαντήσει ε, για το πώ θα λειτουργήσει αυτό. Και η κρατική προεδρία είπε ότι θα προτείνει διάφορα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα νησιά. Θα εργαστούμε και εργαζόμαστε ήδη με τα νησιά και για το ανεπίσημο συμβούλιο να δούμε πώς μπορούν να μπουν στο επίκεντρο των συζητήσεων οι νησιωτικές περιοχές και ε, ο κύριος Αλφόνσε έχει προτείνει τη δημιουργία ομάδα εργασίας και εμείς διαχειριζόμαστε εδώ και καιρό ε, την ομάδα εργασία αυτή. Αυτό για να σας καταδείξουμε ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλά κάπως θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις ανάγκες τους. Θα μπορέσουμε λοιπόν να τα κάνουμε αυτά σε ό,τι αφορά την απόφαση για όλο το νομοθετικό πακέτο, γιατί εδώ πέρα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που αναφέρονται στη συνθήκη. Η περιφερειακή λοιπόν ε, ε, και η ταφική συνοχή δεν είναι κάτι το οποίο αναφέρεται έτσι απλά και γενικά. Το διευκρινίζει, κατοχυρώνεται στην συνθήκη και θα ε, συμπεριληφθεί στο νομοθετικό πακέτο και θα καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εδώ όλοι οι εκπρόσωποι και συναντηθήκαμε χτες μαζί τους, να κάνουμε και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση για τα νησιά. Έχουμε τόσε και τόσε ανακοινώσει για τις, ε, την ύπεθρο, τι ε, νορικέ περιοχέ, ε, τι αστικέ περιοχέ. Μα τα νησιά είναι επίση μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένε ανάγκε. Είναι σημαντικό λοιπόν να το θίξουμε το θέμα αυτό με κάποιο τρόπο και να προσθεθεί αυτό στις διαπραγματεύσεις στη διαδικασία συναπόφαση. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό και όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σα για να κάνουμε σχετικέ συζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινά τώρα η συζήτηση. Συνάδελφο Κοντζόλη έχει το λόγο. Εντάχει, απλώ για να σας χαιρετήσω και να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν απολογισμό σε σχέση με το ταμείο αυτό. Χρειάζεται μεγάλη κινητικότητα. Ε, δεν πρόκειται για μία αντιπαράθεση που έχει διαθεσμικό χαρακτήρα. Η απόφαση είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τις προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί είμαστε φιλόδοξοι, αλλά έχουμε περιορισμένους πόρους και δυστυχώς δεν μπορούμε να προωθήσουμε τις αναγκαίες δράσεις για να προωθήσουμε αυτές τις φιλοδοξίες. Το ζήτημα κατέστη απόλυτα σαφές πρώτα με την Επίτροπο και μετά με τον Κροάτι Υπουργό. Δηλαδή μιλάμε για μια πολιτική ε, συνοχής που αναθέτουμε σε κανονισμούς σε συγκεκριμένους κανονισμούς και στο τέλος τη ημέρας έχουμε ελάχιστους πόρους. Ε, δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε μία μάχη χωρίς όπλα. Μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να καταρτήσουμε το νέο προϋπολογισμό, τους νέους κανονισμούς και μιλάμε για το 1 ή 1,01%. Με τις δυσκολίες έξωθεν ε, σε σχέση με τις νέες μορφές ε, φορολόγησης. Είδατε τι είπε και ο Τραμπ στο Νταβός και ακόμα και ως προς το θέμα της φορολόγησης υπάρχουν, υπάρχουν εν μέρη σύμπνοιες, αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μία συμφωνία. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να κινητοποιηθούμε. Αυτός είναι κρίσιμος χρόνος. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στο διαθεσμικό διάλογο, αλλά να δούμε τις εδαφικές οντότητες, τις περιφέρειες, τις κοινωνικές δυνάμεις. Διαφορετικά εδώ πλέον δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν θα τα καταφέρουμε διότι πολλά λέμε, αλλά δυστυχώς δεν ακολουθούν πράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Στεφάν Μπίζου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και στους δυο σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Όλοι γνωρίζουμε τη τεράστια σημασία που έχει η δουλειά σας, το έργο σας. Θα ήθελα να μιλήσω για το νόημα των πραγμάτων που κάνουμε και για το νόημα των λέξεων γενικότερα. Διάσκεψη παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης. Και εδώ στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το άρθρο 349 που λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Και εδώ έχουμε την έννοια της περιφέρειας. Και επειδή οι λέξεις νοηματοδοτούνται, Οφείλω να σας πω ότι η φύση και το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε μας επιβάλλουν να ε, προβληματιστούμε για την έννοια του τι εστί η περιφέρεια, για την έννοια του τι σημαίνει περιφερειακός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας το οποίο αποτελεί και το βασικό διακύβευμα. Δεν πρέπει λοιπόν να δεχθούμε να είμαστε στη περιφέρεια αλλά να είμαστε στο κέντρο. Οι περιφέρειές μας να είναι στο κέντρο και στο επίκεντρο για εμάς, για τα παιδιά μας και για το μέλλον. Διότι κάθε λέξη έχει νόημα, έχει σημασία. Και από τη στιγμή που γίνεται λόγος για τη λέξη ωκεανός, ας εξελίξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τα πράγματα. Υπάρχουν οι ωκεανοί, αλλά αν δει κανείς ένα χάρτη από το βορρά ή από το νότο, βλέπει ότι κάποια στιγμή ο ένας ωκεανός συναντά τον άλλον. Και μέσα στη λέξη ωκεανός υπάρχει η απεραντότητα αυτού. Και άρα ο μεγάλος αγώνας που πρέπει να δώσουμε για την προστασία αυτού, της απέραντης θάλασσας, στην οποία βρίσκονται τα νησιά μας, τα οποία είναι και στην πρώτη γραμμή που υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε την τεράστια μάχη για την ε, διατήρηση και επιβίωση των ωκεανών γιατί αυτή είναι και ε, η ελπίδα μας για την διάσωση του κλίματος. Έχει υποθεί ότι ο Αμαζόνιος και διάφορα άλλα τροπικά δάση είναι οι πνεύμονες της ανθρωπότητας και ισχύει, αλλά πνεύμονας της ανθρωπότητας είναι και ο ωκεανός και τα ύδατα και οι θάλασσες γιατί ε, προσλαμβάνουν και δεσμεύουν το διοξίδιο του άνθρακα ε, και σε αυτή τη νέα πράσινη συμφωνία πρέπει να έχουμε και τη νέα γαλάζια συμφωνία, Blue Deal, και να δώσουμε στον ωκεανό και στα ύδατα τη σημασία που τους αξίζει. Ο πρόεδρος Μακχούν είπε πριν από δύο εβδομάδες ότι ο ωκεανός αποτελεί κοινό αγαθό της ανθρωπότητας και πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Και επειδή γίνεται λόγος για συνοχή και η λέξη συνοχή έχει και αυτή τη δική της σημασία, θέλω να απευθύνω έκκληση για την εμπειρογνωμοσύνη σας, να τη δεχθούμε, να τη λάβουμε τις εμπειρίες, τις βαθιές σας γνώσεις, διότι ε, ξέρετε το να ε, είναι κανείς σε συνοχή, τι σημαίνει συνοχή, σημαίνει να είναι μαζί ε, και μαζί λοιπόν πρέπει να πορευτούμε, να προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σημερίζομαι την αισιοδοξία σας, μαζί θα προχωρήσουμε και μαζί θα αποδείξουμε ότι οι νησιωτικές περιοχές και οι παράκτιες περιφέρειες είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Στεφάν, λέει ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας, η οποία νοηματοδότησε ε, με ε, πολύ πλούσιες ένδιες στη συζήτηση και είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα συμβάλλει σε όλα αυτά, ε, γιατί όλα αυτά τα οποία μας είπες είναι απαραίτητα επιχειρήματα, ε, απολύτως έγκυρα και έρχονται σε μια έγκαιρη χρονική στιγμή και πολύ τους πιο αξιόμαχα ε, και πιο άξια από τα τεχνικά επιχειρήματα που προβάλλονται ε, στις ε, κατατόπους συνεδριάσεις για τα σχετικά τεχνικά θέματα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Κουταγιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους αλλά και εσάς τους δύο προσκεκλημένους εδώ στην Επιτροπή μας. Αξιολογώ και εκτιμώ ιδιαίτερο στη δουλειά σας και εγώ προέρχομαι από νησιωτική ε, περιοχή, είμαι από την Ίσο Γκότζο, Γκόζο της Μάλτας και ε, ξέρω πόσο πολύ έχετε δουλέψει για να αναδείξετε τις ανισότητες που δυστυχώς επικρατούν μεταξύ των διαφέρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβασα το μανιφέστο το οποίο υπογράψατε στη διάσκεψή σας στο Παλέρμο τον περασμένο Οκτώβριο. Ζητάτε μία μακροχρόνια, μακρόπνοη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να σχεδιάζονται οι αντίστοιχες πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των διαφόρων περιφερειών ε, ώστε να έχουμε ε, ουδετερότητα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό αποτύπωμα ε, με ισορροπημένο τρόπο καθ' όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και τα επόμενα χρόνια, από το 2020 δηλαδή από φέτος και του χρόνου και μετά, στο συντομότερο δυνατό. Συμφωνώ και συμφωνώ και με τους συναδέλφους. Τα νησιά και δεί τα μικρότερα είναι εξαιρετικά σημαντικά όποιο σενάριο και αν επικρατήσει. Και πράγματι πρέπει να τα βάλουμε στο επίκεντρο, ώστε η μετάβασή του σε μια οικονομία δίκαιη με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα ε, να γίνει με ε, φιλικό τρόπο, με ε, όσο τον πιο ουδέτερο τρόπο σε ό,τι αφορά τον αρνητικό αντίκτυπο. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα βελτιώσετε το υφιστάμενο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, ώστε οι οικονομίες μικρότερων κρατών μελών και δινησιωτικών περιοχών να μπορέσουν να ανταγωνιστούν ή, εν πάση περιπτώσει, να μην ε, είναι σε τόσο μεγάλη οπισθοχώρηση σε σχέση με τις κεντρικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ που είστε εδώ. Είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε στενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια Ιζαμπέλ, παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τη διάσκεψη των παρακτήρων περιφερειών της Ευρώπης που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση των σχέσεων σε επίπεδο περιφερειών και φυσικά ε, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφέρειες και τους πολίτες τους και θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τις εργασίες του δόκτωρα Βάσκο Κορντέιρο, του Προέδρου της CPMR. Όπως ξέρετε, δημιουργήθηκε μία ομάδα εργασίας για το νομοθετικό πακέτο 1421 και αυτή η ομάδα που έφερε το όνομα CORE ε, έλαβε υπόψη τα μέλη και τις θέσεις τους ε, της διάσκεψης έτσι ώστε να μιλήσουμε για την πολιτική συνοχής. Για το μετά το 2020 η ομάδα ΚΟΡ και με τα δικά σας αποτελέσματα ζητά την ενισχυμένη υποστήριξη των περιφερειών καθώς και την ε, απλοποίηση της πολιτικής. Πώς ε, είναι δυνατόν ε, η διάσκεψη να βοηθήσει στην επιτέλεση αυτών των στόχων και επίσης ποια είναι η θέση της διάσκεψης σε σχέση με, τους, με τις περιφερειακές περικοπές που ζήτησε ιδιαίτερα το Συμβούλιο και πώς μπορείτε να επηρεάσετε την κατάσταση έτσι ώστε να μην ληφθούν αποφάσεις που αντιτίθενται στα ε, δεδομένα και στους στόχους της διάσκεψης. Ευχαριστώ η Ελιζαμπέτα Κολμίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ τον πρόεδρο Ρώση για την παρουσία του και γιατί μας μίλησε για τις δραστηριότητες της σημαντικής αυτής διάσκεψης όπου συμμετέχουν εκατομμύρια πολιτών. Σημερίζομαι το περιεχόμενο αλλά και το πνεύμα αυτής της πρότασης και θα ήθελα να πω ότι σημεριζόμαστε ε, απόλυτα τις ανησυχίες σε σχέση με τις ενδεχόμενες περικοπές στην πολιτική συνοχής και επειδή το νέο ταμείο το οποίο θα προβάλλει προτάσεις δυνάμει της θέσεις της Επιτροπής, της Ursula von και της ε, πολιτικής συνοχής αφορά ένα 7,5%. Εμείς θα έχουμε 364 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πολύ περιορισμένους πόρους και έτσι με αυτά τα πενιχρά μέσα μπαίνουμε στις διαπραγματεύσεις στο πι χωρίς επιπρόσθετους πόρους. Δηλαδή μειώνονται η πόροι και έχουμε έναν επαρκές ταμείο δίκαιης μετάβασης. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στην αρχική πρόταση που προβλέπεται από το, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 311 της συνθήκης λέει ότι οι πολιτικές πρέπει να ε, την χάνουν χρηματοδότησης από πόρους ε, καθαρά ευρωπαϊκούς, δηλαδή από τους ίδιους πόρους. Αν θέλουμε να φτάσουμε λοιπόν στο νέο πράσινο σύμφωνα ή να προσδώσουμε σημασία στο κοινωνικό πυλώνα, θα πρέπει να μιλάμε για πολιτική συνοχή που αφορούν την συνοχή των περιφερειών μας, δηλαδή να αναθεωρήσουμε τους ίδιους πόρους και να τους συνδέσουμε με νέα έσοδα είτε πρόκειται για το ψηφιακό τομέα είτε τον επιχειρηματικό, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πώς μπορείτε να ενισχύσετε αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με επιπρόσθετους πόρους. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά είναι τα ερωτήματα. Πολύ εμπλουτισμένη η συζήτηση. Πολλές ερωτήσεις μας αφορούν ε, ιδιαίτερως ε, και είδατε ότι επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά γιατί εμείς είμαστε συνομοθέτες και καλούμε να διαδραματίσουμε το ρόλο που μας αναλογεί στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έχουμε την ευθύνη να ε, τροποποιήσουμε τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι έχει να κάνει το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Θα ε, αναλύσουμε προσεκτικά και ελπίζουμε ότι από την ομοπαρασκευαστική διαδικασία θα υπάρξει ένα ταμείο για δίκαιη μετάβαση το οποίο ε, θα έχει διαμορφωθεί με ακόμα πιο δίκαιο τρόπο. Αυτός είναι ο στόχος μας άλλωστε. Πολλά τα ερωτήματα που σας τέθηκαν Σας ευχαριστώ ε, το Μαριάνο και την Ελένη που υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η αρχή της εταιρικής σχέσης, την οποία ήθελε και να αμφισβητήσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και μπορέσαμε σε αυτό το στάδιο με την ε, προσωρινή ε, ε, κοινή ε, ε, κατανόηση και συνένεση να διατηρήσουμε αυτή τη διαπίστωση και αυτή την αρχή. Το πρόβλημα αυτό τίθεται και στο πλαίσιο του Interreg, το οποίο γνωρίζω καλά γιατί αφορά και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αφορούσε ε, πριν γίνει η τροποποίηση στην τελευταία διαπραγμάτευση. Σήμερα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με τα νησιά και το Interreg. Υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει θέμα. Άρα εμείς έχουμε την εξής αρχή. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία επί όλων των θεμάτων, δεν υπάρχει συμφωνία επιμέρους ε, για κάποιο θέμα. Δεν υπάρχει συμφωνία για τίποτα μέχρι ότου υπάρχει συμφωνία για όλα. Έχουμε εισηγητή για το θέμα αυτό, το Πασκάλ, και θα... Ε, βγούμε από αυτή τη διαπραγμάτευση έχοντας λύσει το θέμα του ίντερεγ και των νησιών ή τουλάχιστον αυτή την ευχή και επιθυμία διατυπώνω να ρυθμιστεί, να μεθοδευτεί ξεκάθαρα το ζήτημα των νησιών και μάλιστα με τον πιο συγκεκριμένο, τον πιο ακριβή ε, τρόπο, τον βέλτιστο δυνατό τρόπο γιατί αν κανείς επαφίεται μόνο στις ε, ερμηνείες ε, των κειμένων έτσι όπως θα προβεί σε αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια σίγουρα αφήνει το δρόμο ανοιχτό για διάφορα προβλήματα. Πασκάλ όμως σας ξέχασα και σας δίνω το λόγο. Φρανσουά, Αλφονσί ίσως, όχι Πασκάλ. Δεν πήρα το λόγο προηγουμένω. Είμαι ο Φρανσουά Αλφονσί και λυπάμαι που δεν το πήρα το λόγο για να χαιρετήσω ε, τον Περιφερειάρχη που είναι πιο κοντά σε εμά, στην Κορσική. Και γεωγραφικά είναι πιο κοντά η Τοσκάνη, αλλά και έχουμε μια ε, ψυχική αδελφοσύνη που μα ενώνει η Κορσική με την Τοσκάνη. Απέναντι είμαστε άλλωστε. Θέλω να χαιρετήσω τον πρόεδρο Ρώση για την παρουσία του εδώ, τον Περιφερειάρχη και Αντιπρόεδρο. Ε, και συμφωνώ απολύτως με τα λόγια του Προέδρου μας, του κυρίου Ομαχζή. Για να είμαστε αποτελεσματικοί και για να μπορούμε να δράσουμε, χρειαζόμαστε ισχυρούς περιφερειάρχες, διότι υπάρχει ανάγκη να δοθεί πολιτικό βάρος στις προτάσεις μας, το απαραίτητο πολιτικό βάρος, το οποίο έχουν ε, πολιτικοί άνδρες και γυναίκες σημαντικοί. Η συνεργασία μας ε, δεν είναι προφανής, ε, δηλαδή υπάρχει αλλά δεν έχει πολλαπλασιαστεί, δεν έχει φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε. Πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερες συναντήσεις. Έχουμε συνομιλητή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να βασιστούμε και στα κράτη-μέλη. Και ξέρετε, οι ευρωβουλευτές ε, συχνά στην χώρα τους, να το πω έτσι δεν περνάει και φοβερά ο λόγος τους ε, όταν επιστρέφει ο Ευρωβουλευτής ε, στη χώρα του. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει μια μέθοδος που μπορεί να μας ε, βοηθήσει. Η διάσκεψη των παράκτων περιφερειών της Ευρώπης είναι εργαλείο για να καλλιεργήσουμε, να ενισχύσουμε τις σχέσεις με τις χώρες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εντείνουμε την πίεση που ασκούμε και άρα να φέρουμε αποτελέσματα. Εντατικοί μήνες θα είναι οι επόμενοι μήνες στους οποίους θα εργαστούμε με πολύ μεγάλη σημασία ε, για το ευίωνο μέλλον των ε, περιφερειών. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Ρώση. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους. Πρόκειται για μια συζήτηση υψηλού επίπεδου που θίγει πληθώρα ερωτημάτων όταν ως πολίτης αλλά και ως θεσμικός άκουσα την κυρία Φοντερ Λάιεν να μιλάει με αποφασιστικό τρόπο για αυτό το πρότυπο, το αναπτυξιακό πρότυπο οικολογικών διαστάσεων, είδα ότι μπορούμε να ε, συνδέσουμε την Ευρώπη με τον πολίτη, να το συμφιλιώσουμε. Ε, για να φτάσουμε σε μία πλήρη ανάπτυξη ε, σε εκθετικό βαθμό. Και αυτός ο δρόμος είναι αποφασιστικής σημασίας για γυναίκες, άνδρες, ολόκληρο τον πλανήτη. Νομίζω ότι η Ευρώπη έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, διότι γνωρίζει ε, ο πολίτης ότι δεν μπορούν να λυθούν περιβαλλοντικά ζητήματα ε, μέσα σε κλειστές πόρτες, στα εθνικά δηλαδή πλαίσια. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τις, ε, τους πόρους που είναι διαθέσιμοι έχουν γίνει όμως ε, περικοπές, περαιτέρω περικοπές σε σχέση με την προηγούμενη επταετία και δυστυχώς θα παλινοδίσουμε. Γυρίζουμε την πλάτη στην Ευρώπη, στην ουσία. Ε, εγώ δέχομαι αυτή την έκκληση, θα την αναφέρω στη διάσκεψη των παρακτήων θαλάσσιων περιοχών για μια κινητικότητα για την οικολογική μετάβαση. Νομίζω ότι τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κινητοποίηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα αποφασιστικής σημασίας ε, σήμερα θα ήθελα να πω στον κύριο Γκουαλμίνη ότι μπορούμε να δεχτούμε τους δείκτες της ομάδας Μόντι που έχουν την αξία ε, να μην βάζουν το χέρι στην τσέπη του φορολογούμενου. Μπορούμε να βρούμε πολλούς πόρους και να δώσουμε και ένα προφίλ ίδιων πόρων εκεί που χρειάζεται. Θα ήθελα να πω σε σχέση με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, νομίζω ότι υποτιμούμε μία πτυχή σημαντική δεν αφορά μόνο τα ορυχεία ή ειδικότερε καταστάσεις, αλλά πολλούς παραγωγικούς τομείς. Στην περιφέρειά μου υπάρχει το ε, θέμα του περάσματος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οποίο σημαίνει ότι θα γίνει μία ε, ολίσθηση στην απασχόληση. Αυτή η μετάβαση είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους τους τομείς. Ο κάθε τομέας θα πρέπει να ε, προβεί, να οδηγηθεί σε συγκεκριμένες ε, ε, μεταλλαγές. Το είδαμε για... και στην περίπτωση των πλαστικών, δηλαδή το γεγονός ότι βάλαμε ένα απειροελάχιστο ποσό ως φορολόγηση στις πλασικές σακούλες οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στο να απομακρυνθούν. Άρα θα πρέπει να ξαναδούμε την αρχή του Just Transition για να φτάσουμε σε εργασία, σε μεγάλες επενδύσεις. Διαφορετικά αυτό το θετικό αίσθημα έναντι της Ευρώπης θα εκλείψει θα πρέπει να δείξουμε ότι πραγματικά δίνουμε μάχη για την οικολογική μετάβαση. Διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε απολύτως τίποτα. Σημερίζομαι αυτή την έκκληση, γι' αυτό υπάρχει και η διάσκεψη μέσα στα πλαίσια του νησιωτικού χαρακτήρα, των παρακτήων περιοχών και ούτω καθεξής, γιατί θα πρέπει να υποστηρίξουμε την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει και με τις ε, δασικές περιοχές. Όσο μεγαλύτερες δασικές περιοχές έχουμε, τόσο απορροφάται το διοξίδιο του άνθρακα. Το ίδιο αφορά και τη θάλασσα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, όλες αυτές τις αλλαγές. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το σκάνι έχει μεγάλη σχέση με την ε, κορσική. Η ιδιόγλωσσα, η διάλεκτος που μιλάμε έχει πολλά στοιχεία της κορσικής και αντίστροφα. Γι' αυτό ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, παντού δημιουργούνται βουνά πλαστικού και θα πρέπει αυτά τα πλαστικά να απομακρυνθούν διαφορετικά μπορούν να ε, θανατωθούν και τα κητοειδή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στις θαλάσσιες περιοχές και στις δασικές εκτάσεις που αποτελούν τον πνεύμονα της γης, έτσι ώστε να μην αποδυναμωθεί αυτό το πλαίσιο δράσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη συνεργασία Interreg και γι' αυτό δώσαμε και μεγάλη μάχη. Τώρα θα ήθελα να εκφράσω μια προσωπική γνώμη ως προς την ανταγωνιστικότητα. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια διαφορετική αιρεσιμότητα σε σχέση με την μακροοικονομική. Η αιρεσιμότητα θα πρέπει να συνδέεται με σχέδια και προγράμματα που υλοποιούνται στις περιφέρειες ή σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να φτάσουμε στην ουδετερότητα ως προς τη χρήση του άνθρακα. Γι' αυτό χρειάζονται προγράμματα δράσης που να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση της ουδετερότητας. Αυτό θα ήταν και η χρυσή τομή και παράλληλα θα είχαμε και την συνδρομή των διαφόρων ταμείων, καθώς και την κρατική συνδρομή που θα είχε επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον, πέρα από τους μηχανισμούς της αγοράς. Αυτά ήθελα να σας πω ευχαριστώντας σας για τη δυνατότητα που μας δώσατε να λάβουμε το λόγο και για την όθηση αυτή, διότι πραγματικά πιστεύετε στο ε, ρόλο των ε, ντόπιων, των εγχώριων θεσμών. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με ε, μια Ευρώπη που κινείται σε επίπεδο διακυβερνητικής ε, πορείας, δηλαδή μιλάμε για μια διακυβερνητικότητα η οποία δεν ξέρω αν αποτελεί και το σωστό σκέλος προώθησης των σχεδίων που επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο συναδελφός μας ο Φρανσουά Αλφονσί, χρειαζόμαστε ε, τους δε. χρειαζόμαστε, σας χρειαζόμαστε πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντική διάσκεψη για τις πρακτικές περιφέρειες της Ευρώπης για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών Περιφερειών τους επόμενους μήνες. Οι έξι μήνες ε, οι επόμενοι θα καθορίσουν ε, τη ζωή των ε, πολιτών στις περιφέρειες αυτές για την επόμενη δεκαετία. Θα πρέπει λοιπόν να μην τους απογοητεύσουμε και να μην ε, ξεχάσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και λέμε μετά ότι α, πρέπει να έχουμε κάνει και αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν που έχουμε την υποστήριξή σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι, ολοκληρώνουμε τη συνεδρίασή μας. Όπως τα γνωρίζετε, η συνεδρίαση των συντονιστών έγινε σήμερα το πρωί και λάβαμε ε, μία σειρά αποφάσεων. Θα σας αποστείλουμε μέσω email. Έχετε ήδη λάβει τα σχετικά email και αποφασίσαμε να κάνουμε μία ανακοίνωση τύπου σε σχέση με την απόφαση που ελήφθησε ομόφωνα από τους συντονιστές σήμερα το πρωί. Θα βρείτε λοιπόν όλα αυτά στα email σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, σημεία στα διάφορα τα οποία θα θέλετε να δείξετε. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο. Η επόμενη συνεδρίαση λοιπόν θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 19 Φεβρουαρίου στις 3 ε, το απόγευμα μέχρι τις 6.30 και στις 20 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλες